Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου ε, προέβη στην διαπίστευση των κυρίων Κορνιγέ και ε, Λαλόντ και αναλαμβάνουν ε, και επίσημα τη θέση από τις 18 Μαΐου. Υπάρχουν